Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε, παρακαλώ. Ε, sorry, silence please. We want to begin because... Θέλουμε να ξεκινήσουμε γιατί θέλουμε να τα κάνουμε τα πράγματα στην ώρα τους. Λοιπόν, Έχετε όλη κάρτα ψηφοφορίας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω ότι χθες έγινε συνεδρίαση των συντονιστών και οι αποφάσεις τους σας αποσταλούν. Ελήφθηκαν πάρα πολλές αποφάσεις, αλλά τελειώσαμε πολύ αργά. Θα λάβετε τις αποφάσεις τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, προτείνω, αντί αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι την Παρασκευή στις 12, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Περνάμε τώρα αμέσως ε, στην ψηφοφορία, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ψηφοφορία. Στις 10 η ώρα θα έρθει ο Επίτροπος Λαβράτσης και στις 2.30 θα φύγουμε για να πάμε ε, στην αποστολή μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσως με τον κατάλογο των ψηφοφοριών και να ξεκινήσουμε με την έκθεση του συναδέλφου Μιρτσέα Διακόνου του Αντιπροέδρου για την πιθανή επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι αυτό το σχέδιο υποβλήθηκε στις 23 Μαρτίου. Υπήρχε προθεσμία στις 30 Μαρτίου για υποβολή τροπολογιών. 137 τροπολογίες. Είχαμε γνωμοδοτήσει τη επιτροπή Τραν και Ρέτζι. Λάβαμε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Είδα ότι έγινε πολύ καλή δουλειά με τις συμβιβαστικέ προτάσεις, αλλά είναι αρκετά μεγάλη ψηφοφορία. Θα ήθελα να ε, ρωτήσω τον συναδελφό Διακόνο αν θέλει να πάρει το λόγο τώρα ή μετά. Όχι, ωραία. Να συνεχίσουμε για να προλάβουμε κιόλας. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 4 της παραγράφου 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία υπεριθμών 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Πρόταση της τραν, τραν 6, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρόταση Ρέτζι 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40, Winkler, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 ντράγκητσι, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα κάνουμε μια επαλήθευση για τη 41. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά προτιμώ να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Α, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία, δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Υπάρχει ένας επιπλέον από τους πρασίνους. Οι πράσινοι έχουν ένα επιπλέον συνάδελφο. Ψηφίσατε. Δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας. Μπορεί κάποιος ε, να το δει. Could you check now? Ah, the next place. Μπορείτε να αλλάξετε θέση. She has to move. Yes. You can move to the other. Μπορείτε να πάτε στη διπλανή θέση καλύτερα. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Allora, il voto ancora per. Ωραία. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σαράντα τρία Ζαγοράκης. Α. Α, με συγχωρείτε, απορρίφθηκε, δεν εγκρίθηκε. Περνάμε σε 42, Μαραγκάλι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43, Ζαγοράκης, υπέρ, κατά, αποχές εκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λιμπάτσκα 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση παρακαλώ, γιατί είναι οριακά τα θέματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiudo la votazione. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Ωραία. Περνάμε στην 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, και εδώ θα κάνουμε μια παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι σαφές νομίζω. Να ξαναδούμε. 56 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Για μία ψήφο. 57. Τραν 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε διάφορες τροπολογίες της Ρέτζη. Ρέτζη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζη 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζη 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζη 9 υπέρ κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Ρέτζι 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 11 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 664 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 67 με προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 15 10 ψήφους υπέρ, 15 κατά. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30-32 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι 333 30-33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία, 73, να τα πάω λίγο πιο αργά. 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Σπίντο. Απορρίπτεται. 74. Ε, 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 75. Συγγνώμη, συγγνώμη. Allora, 76... Ε, 76 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 με προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 με προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την τραν 16. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 με προφορική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε, διότι δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 90. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά. Υπέρ, συγγνώμη, ποιος είναι, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη. 95 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 με προφορική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 αποσύρθηκε 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 με προφορική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται είναι ταυτόσιμη με την 112, επομένως εγκρίνεται και οι δύο και περνάμε στην 113, Μαλτέζε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 17, 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 με την προφορική τροποποίηση 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 πως τροποποιήθηκε με την προφορική τροποποίηση τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 8 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά απορρίπτεται με μία ψήφο 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 19. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για την Τραν 14. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Ετράν τραν 19 υπέρ κατά αποχές το, το χέρι σας να σηκώνετε παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 28 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τραν 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 31. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, ένα ψηφοφορίας. Λήξη ψηφοφορίας. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν περισσότερε ψήφοι κατά, αλλά μάλλον έκανα λάθο. Ρέτζι 2. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Ρέτζι 3. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Ρέτζι 4. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Ρέτζι 5. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 9 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 135. Καρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 138. Βέντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140. Χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές. Πρώτο τμήμα. Για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα έναρξη ψηφοφορίας λήξη ψηφοφορίας συγγνώμη Νόμιζα ότι η ομάδα σας είχε σηκώσει το χέρι στο κατά. Μπορεί να, το, να, να είδα λάθος. Με συγχωρείτε. Ε, δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 140. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 2 υπέρ κατά αποχέ κατά κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 3 Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το τραν 2. Ε, ενα ψηφοφορίας. Close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, δεν το έθεσα σε ψηφοφορία γιατί ήταν σαφέ, λέει η πρόεδρο. Τραν 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το τραν 4. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Είναι μικρή διαφορά, γι' αυτό πολλές φορές δυσκολεύομαι. Τραν 5. Υπέρ, κατά, αποχές. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τραν 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Είδατε με πολύ μικρή διαφορά. Τραν 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να προσθέσουμε άλλη μία που δεν υπάρχει στον κατάλογο, άλλη μία τροπολογία, την Τραν 39. Δεν είναι στον κατάλογό σας. Ο εισηγητής είναι κατά. Το θέτω στην ψηφοφορία τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 11. Συγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 152, Βίνκλερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 Βίνκλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 158, Κρασνοντεύσκη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 159 με, την προφορική τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 12 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πάμε στην συμβαστική πρόταση 13 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τραν 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ένα ψηφοφορίας για την 168 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 8 Ζαγοράκης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε. Για την τροπολογία 10 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορίας. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 17 ψήφου υπέρ. Ε, τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 να το επαληθεύσουμε. Για το 13 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά όμως, να το τονίσω αυτό. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη Β, υπέρ, εγκρίνεται. 17, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση του συζητητή Παριθμόν 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία 22, Κρασνοντεύσκη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 27, Κρασνοντεύσκη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 Μαραγκάλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 Νέκοφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, την παραπομπή 4 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 Βίνκλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης στο σύνολό της. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Bene, complimenti al relatore, 22... Συγχαρητήρια στον εισηγητή, 22 ψήφοι υπέρ, καμία Κατά και δύο εποχές. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν στον συνάδελφο Διακόνους. Ευχαριστούμε τους και όδης και τη Γραμματεία για την πολύτιμη βοήθειά τους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση. Να ακούσουμε τον κύριο Διακόνου να μας πει δύο λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη που καθυστέρησα να ανάψω το μικρόφωνο μου. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τις πολλές τροπολογίες και για τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Αυτό όμως δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα. Και άρα, όχι, ε, δεν σας ζητώ μόνο συγγνώμη, αλλά σας ευχαριστώ και θερμότατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. E Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά. Πρόκειται για μια πλούσια έκθεση. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη έκθεση που θα ψηφίσουμε. Πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότηση του Μπόγκταν Ντροβιέσκη για την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2016. Ε, γνωρίζετε ότι υπευλήθηκε το, στις 4 Μαΐου, προθεσμία κατάθεση τροπολογίων 12 Μαΐου και υπευλήθησαν 30 τροπολογίες. Γνωρίζετε μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ε, να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για την συνεισφορά της Επιτροπής Προπολογισμού για τη διαπραγματευτική εντολή που θα εγκριθεί στη συνέχεια από την Ολομέλεια τον Ιούλιο. Θέλει να πει ο συνάδελφος κάτι? Όχι, ωραία να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11. Ε, κατά τμήματα, Εσεντή το ζήτησε. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ίσως απορρίπτεται ίσως εγκρίνεται αλλά εμπασευτός να το ελέγξουμε να το επαληθεύσουμε ξεκινάει η ψηφοφορία το δεύτερο τμήμα της 11 ψηφίζουμε πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 12 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Τροπολογία 21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Με την προφορική τροπολογία της Πέτρα Καμερέβερτ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην παράγραφο στην συμβαστική τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τρίπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 Θέλετε να ελέγξουμε τη 2 Ανοίγει η ψηφοφορία για την, ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη Α, τροπολογία 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη 3, Λουίτζι Μόργανο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ξεκινάει η ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρας της ψηφοφορίας. Πολύ γρήγορα πάμε, πώς, όχι. Καλώς. Συγχαρητήρια. Στο συνάδελφο Δρογκεύσκη, 21 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, γεγονός που ενθαρρύνει τον εισηγητή μας να προχωρήσει με τον προπολογισμό. Να περάσουμε τώρα στην τελευταία ε, έκθεση που έχουμε προς, έκθεση, ε, προς ψήφιση, την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Διακόνου Να την προσθέσουμε γιατί δεν ψήφισε. Να προσθέσουμε μία ψήφο υπέρ της ε, συναδέλφου Ζιντρόβα για την προηγούμενη έκθεση, την τελευταία ψηφοφορία. Και περνάμε τώρα στην πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα. Είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Διακόνου, η οποία δεν είναι σήμερα, του κυρίου Διακόνου, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ, γιατί σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ε, συνεδριάσεις. Ξεκινούμε με την πρώτη τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 του εισηγητή, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 τροπολογία, νέκοφ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Πατρίσια Πατρίσιαλο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, κατά, αποχές, Ίσως εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία δια της ηλεκτρονικής οδού πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Διορθώνω. 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 ψηφοφορία κατά τμήματα ζητά το ΕΛΚ. Το πρώτο τμήμα της 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 30 ζουλό. Υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 2 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 φορική τροπολογία Νέκοβ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται.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 Ξαναψηφίζουμε παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορία. 23... 23 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ε, πολύ σημαντική επιτυχία. Κύριε Διακόνου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ε, Δώστε ένα μικρόφωνο στον Αντιπρόεδρο Διακόνου. όταν αποφάσισα να υπερασπιστώ αυτό το θέμα στην Επιτροπή του Πολιτισμού και να το αναλάβω. Ήταν πολύ λίγοι παρόντες και σας είχα τότε ε, παρουσιάσει ένα αντικείμενο που είχε κατασκευαστεί στο Δέλτα του Δούναβη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ψηφοφορία. και θα σας στείλω τέτοιου είδους αντικειμένα στον καθένα σας. Ευχαριστώ θερμά. Ωραία. Έχουμε και την εκπληξούλα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε να δούμε τι άλλα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης συγκεκριμένης έχετε να μας δώσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Είμαστε στην ώρα μας ε, ακριβώς σήμερα. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν ε, του Επιτρόπου Νταβράζης. Τα, να κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα λοιπόν μέχρι να έρθει ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Welcome, Καλώς ορίσατε αγαπητέ Επίτροπε. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που η Επιτροπή μας έχει την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί σας και να ακούσει η Επιτροπή μας τις προτάσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις γραμμές της πολιτικής για θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά που αφορούν και την νεολαία. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά, αν μου επιτρέπετε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο Επίτροπος, ε, φυσικά, και βεβαίως θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα, την οποία θα θέλαμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε, να έχουμε ε, συνεχείς ε, επαφές, ε, να μην έχουμε απλώς τυχαίες συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως και του Συμβουλίου. Γνωρίζετε ότι προσπαθούμε να έχουμε μια νέα εποχή διοργανικών σχέσεων και επομένως θεωρούμε ότι αυτή η σχέση πρέπει να ενισχυθεί για να έχουμε και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και δυνατότητα συνεργασίας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για το Συμβούλιο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε πληροφορίες και ε, στην εξέλιξη των προγραμμάτων. Εμάς μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα προγράμματα που αφορούν ε, το φακελό σας, ε, το Erasmus το πρόγραμμα για τις ε, πολιτικές της νεολαίας και θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο του προγράμματος Juncker. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Επομένως, θα υπάρχει χρόνος για να ακούσουμε εσά για 10 λεπτά περίπου στην αρχή και από εκεί και πέρα να ακούσουμε παρεμβάσεις, να συλλέξουμε ερωτήσεις και να δοθούν και κάποιες ε, απαντήσεις θα ήθελα να επισημάνω τρία ζητήματα τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Καταρχάς ε, υπάρχει μια ανησυχία της Επιτροπής μας. Μόλις δόθηκε εντολή για τον ε, ε, προϋπολογισμό στον συνάδελφο Ζωβιέσκη, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας, για τον τριμερή διάλογο και για να προχωρήσουμε για τον προπολογισμό του 2016. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στα πολιετά ε, προγράμματα είχαμε μια σημαντική αύξηση του προπολογισμού για το Εράσμους και για τη Δημιουργική Ευρώπη, ενώ υπήρξε μείωση στον προπολογισμό για άλλε πρωτοβουλίε και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Παραδείγματο χάρη κάποια πιλωτικά προγράμματα, στα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει ε, μειωμένο προπολογισμό. Ε, ελπίζουμε να μπορούσουμε να βασιστούμε και στη δέσμευσή σας για να προχωρήσει ο προπολογισμό του 2016 και να τον αυξήσουμε κιόλας ε, διότι είναι αλήθεια ότι θα υπάρχει αύξηση του προπολογισμού για την ε, δημιουργική Ευρώπη, αλλά για το 2016 υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες θέλουν να μειώσουν το συνολικό ποσό. Ε, βραβεία τύπου Μελίνα Μερκούρη, ε, βραβεία για τον πολιτισμό, τα οποία ε, θα μειώσουν τελικά το συνολικό ποσό. Υπάρχουν επίσης και οι πληρωμές πέραν από τις επενδύσεις, ε, το συζητήσαμε και χθε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν και την άποψή σας επ' αυτού και θα θέλαμε ε, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Να πω κάτι γενικό και από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι θα σταθούν σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Εμάς μας ανησυχεί και ένα άλλο θέμα, πιο πολιτικό. Στα δέκα σημεία του προγράμματος Juncker το θέμα πολιτισμός και παιδεία σχεδόν δεν εμφανίζεται καθόλου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που αποτελεί οπισθοδρόμηση και σε σχέση με την Ευρώπη 2020 και για το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, επανεξετάσουμε τη στρατηγική ε, εκπαίδευση 2020 ε, και θα ήθελα να ξέρω και τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς και η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού για να μπορέσουμε να έχουμε πιο προβεβλημένα ε, στις προτεραιότητες αυτές του προγράμματος Juncker τα θέματα του πολιτισμού, της δημιουργικότητας, ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, μόλις εγκρίθηκε και μία έκθεση της Επιτροπής μας για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πολιτιστικών θεμάτων αλλά και για θέματα παιδείας. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι επ' αυτού δεν είναι κατάλληλη η προσοχή που δίνεται στα θέματα. Γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχει καν κοινωνική ένταξη ε, και ευφυής ένταξη εάν ε, ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικά συστήματα πολλών ε, χωρών, και ευρωπαϊκή κινητικότητα σπουδαστών και φοιτητών και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και επένδυση στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Για μας είναι ουσιαστικό ζήτημα και πρέπει κάποιος να μας διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν αυτά. Όσον αφορά το σχέδιο επενδύσεων Juncker, σίγουρα θα το θίξουν και οι συνάδελφοι. Το 2016 θα υπάρχει αυτή η καινοτομία, αυτή η σημαντική ευκαιρία, η οποία όμως δεν ξέρουμε αν περιλαμβάνεται το θέμα της παιδείας. Τι ε, προγράμματα και τι πλατφόρμες σκοπεύετε να προωθήσετε σε θέματα παιδείας ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Connect. γιατί ε, κάναμε ένα κοινό σεμινάριο για να δούμε τι προοπτικές έχουμε για το e-learning και το e-teaching κυρίως. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες επενδύσεις στην παιδεία και σε εκπαιδευτικές υποδομές. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, ε, βιομηχανίας πολιτισμού και δημιουργικότητας, ε, το οποίο συμπεριλέβεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν υπήρχε αρχικό στο πρόγραμμα Juncker. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν μια διαβοβαίωση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά, να ξέρουμε ότι έχουν συμπεριληφθεί. Επίσης θα θέλω να μου πείτε τι κάνετε εσείς μαζί με τον συνάδελφό σας τον κύριο Έτιγκερ για τα όλα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργικότητα, τα οπτικοακουστικά μέσα και επίσης τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στον πολιτισμό ε, εντός της ε, πρόκλησης της ψηφιακής αγοράς. Αυτά σας τα παρουσιάζω ως μια εικόνα των θεμάτων που μας απασχολούν. Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι με τις ερωτήσεις τους θα διευκρινίσουν λίγο καλύτερα τι ακριβώς θέλουν να ξέρουν. Σήμερα το απόγευμα θα επισκεφτούμε μαζί την υπηρεσία ε, ΕΑΣΑ ε, και θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα με διάφανο τρόπο και γι' αυτό είμαστε βέβαιοι με ποιο τρόπο εφαρμόζονται τα διάφορα προγράμματα και ε, κατά πόσον γίνονται σεβαστές και οι διατάξεις που έχουμε συμπεριλάβει στους κανονισμούς. Ε, κάποιες φορές έχουμε κάποιε ανησυχίε και σήμερα η επίσκεψη αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς προχωρούν τα θέματα. Ε, θα σας δώσω αμέσω το λόγο, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σα παρουσία και από εδώ και, και πέρα θα δοθεί ο λόγο στους συναδέλφου. Παρακαλώ κύριε Πίτρο. Thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Την τελευταία ευκαιρία που είχα να έρθω εδώ, πριν από ένα μήνα περίπου, μιλήσαμε για ευρεία, για οριζόντια ζητήματα. Είχαμε την πρώτη συζήτηση για το πεδίο αρμοδιοτήτων μας και σήμερα έχουμε πλέον την ευκαιρία να μην μιλήσουμε γενικά, αλλά να μπούμε σε λεπτομέρειες. Να εμβαθύνουμε. Καταρχάς, να σας αναφέρω τρεις από τις προτεραιότητές μου, που έχουν να κάνουν κυρίως με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Γιατί πολλά έχουν συμβεί το περασμένο μήνα ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις και θα υπάρχουν και νέες εξελίξεις που μπορούν ε, να επηρεάσουν τα της ε, εκπαίδευσης τους επόμενους μήνες. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η παιδεία ορίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πολιτική που υπόκειται στην πολιτική απασχόλησης. Επομένως, βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει στις διαδικασίες και στις διεργασίες η εκπαίδευση που θα προωθήσουν την απασχολησιμότητα που θα βοηθήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διεργασίες και οι διαδικασίες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έτσι ώστε οι φοιτητές, μαθητές και λοιποί να είναι περισσότερο απασχολήσιμοι στην αγορά εργασίας. Είναι ένα σημαντικό φαινόμενο αυτό και είναι μια καθοριστική στιγμή, η στιγμή κατά την οποία πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υπάρχει ακόμα περισσότερη απασχολησιμότητα. Έχουμε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και οι βασικοί τίτλοι, οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές εκεί είναι σταθεροί. Στην εκπαιδευτική πολιτική μπορούμε να πούμε ότι πλησιάζουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική Ευρώπη για το 2020 και αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλη πιθανότητα πράγματι να τους καταφέρουμε, να τους πετύχουμε τους στόχους αυτούς μέχρι το 2020. Όμως η απασχολησιμότητα και το να γίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο αποτελεσματικά είναι βασικό στοιχείο του διαλόγου που έχουμε εμείς με τα Υπουργεία Παιδείας των κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά, τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες τραγικών γεγονότων στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές κοινωνίες. Σας υπενθυμίζω ότι συνέβη στο Παρίσι, στην Κοπενχάγη και στις Βρυξέλλες, όπου νέοι εξτρεμιστές επιτέθηκαν σε πολίτες, κάτι το οποίο καταδεικνύει ότι λείπει ένα βασικό στοιχείο ή έχει αποδυναμωθεί ένα ε, ουσιαστικό στοιχείο των κοινωνιών μας. Και αυτό το κάτι είναι η δημοκρατική κοινωνικοποίηση. Επομένως, το νέο φαινόμενο στην εκπαιδευτική πολιτική, στον εκπαιδευτικό τομέα, είναι ότι πρέπει να διερευνήσουμε ε, ποια στοιχεία είναι αυτά που αποδυνάμωσαν τη δημόσια εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Πού είναι οι ρίζες αυτής της διαδικασίας αποξένωσης και αλωτρίωσης ε, των συγκεκριμένων νέων ανθρώπων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τον εξτρεμισμό και τον ρίζοσπαστισμό στις δημοκρατικές κοινωνίες. Και βέβαια τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα σχολεία και οι δάσκαλοι είναι στοιχεία κλειδιά σε αυτή τη διαδικασία. Τα σχολεία και οι δάσκαλοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επιτυγχάνουν τη δημοκρατική κοινωνικοποίηση, μπορούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις δημοκρατικές αξίες, μπορούν να διδάξουν στους λαούς τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα κάνουν τους μαθητές να ε, μπορέσουν να ταιριάξουν στην ευρεία κοινωνία και να νιώθουν άνετα με τις αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας. Γι' αυτό και εμείς μαζί με ε, το Γάλλο και τον ε, Λετονό Υπουργό Παιδείας μετά από τις επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπενχάγη έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία την οποία αποκαλούμε διαδικασία μετά το Παρίσι έναν διάλογο πολιτικής με τους Υπουργούς Παιδείας. τον ξεκινήσαμε στο Παρίσι ε, στις 17 Μαρτίου με στόχο να αναβαθμίσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να γίνει ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα σχολεία, οι δάσκαλοι μπορούν να προωθήσουν τη δημοκρατική κοινωνικοποίηση, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εξτρεμισμό στους νέους και πώς μπορούν οι Υπουργοί Εκπαιδευτικής Πολιτικής να συνεργαστούν για την ενίσχυση δημοκρατικών αξιών, για την ενίσχυση της έννοιας του πολίτη ε, στα προγράμματα σπουδών των σχολείων. Όπως σας είπα, αυτή η διαδικασία ε, ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου. Το Μάιο έγινε το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών όπου συζητήθηκαν οι νέες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα γιατί η επικείμενη Λουξεμβούργια Προεδρία, Προεδρία του Λουξεμβούργου, έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και έχουμε μεγάλες πιθανότητες να καταφέρουμε να εγκριθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του 2015. Τώρα, βασικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας είναι για να σας δώσω κάποια παραδείγματα να δοθούν παραδείγματα στα εκπαιδευτικά συστήματα και να έχουμε κάποιες ε, θεμέλιες λίθους να το πω έτσι έτσι ώστε τα σχολεία να αναπτύξουν τέτοιου είδους δεξιότητες τους μαθητές τους δηλαδή να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος, να προωθηθεί περισσότερο ε, η δυνατότητα ανάγνωσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας ε, μεταξύ άλλων. Αρμοδιότητα δικιά μου είναι να προωθήσουμε να βοηθήσουμε τα Υπουργεία Παιδείας ε, των κρατών μελών ή ε, τα περιφερειακά ε, Υπουργεία Παιδείας όταν μιλούμε για χώρες που είναι ομοσπονδιακές ε, έτσι ώστε τα Υπουργεία να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες αυτές που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία και πανεπιστήμια για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και της δημοκρατικής κοινωνικοποίησης. Το δεύτερο στοιχείο που είναι απαραίτητο και σημαντικό ως εξέλιξη είναι το εξής περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εξωτερικών σχέσεων και της πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής και των προτεραιοτήτων της πολιτικής γειτονίας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα η δική μου Γενική Διεύθυνση πλησίασε την Αντιπρόεδρο ε, και την ε, ύπατη εκπρόσωπο ε, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έτσι ώστε η διάσταση του πολιτισμού των αθλημάτων να, μεταξύ άλλων να συμπεριληφθεί στην πολιτική εξωτερικών σχέσεων. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη είναι η πιο ισχυρή στον κόσμο. Γιατί, γιατί η Ευρώπη δεν έχει δικό της στρατό, δεν έχει μία αστυνομική δύναμη, έχει όμως μία ευρωπαϊκή κουλτούρα, έχει την εκπαίδευση, την παιδεία, τα αθλήματα, όλα αυτά τα τεράστια επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι σημείο αναφοράς παντού στον κόσμο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα είναι καλά παραδείγματα για ε, τα άλλα έθνη, τις άλλες περιοχές και βλέπουμε ότι τα αθλήματα, ο αθλητισμός χρησιμεύει ιδιαιτέρως για να προωθήσει τα ιδανικά, τα ιδεώδη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Με χαρά μου λέω ότι η Αντιπρόεδρος ε, και το γραφείο της και ο αρμόδιος επίτροπος για την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, συνεργάστηκαν μαζί μας πολύ επικοδομητικά και άρα έχουμε πολλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε, δηλαδή να ε, θεσμοθετήσουμε κάποια βασικά στοιχεία πολιτιστικής και πολιτισμικής διπλωματίας που θα αποτελέσει μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω βέβαια τη σημασία της αρχής της επικουρικότητας. Δεν θέλουμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ένα υπερεθνικό επίπεδο πολιτιστικής και πολιτισμικής δράσης. Δεν έχω καμία πρόθεση να είμαι ένας υπερυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μόνο που θέλω είναι να προωθήσω, να βοηθήσω, να συντονίσω ε, τις προσπάθειες των κρατών μελών. Υπάρχουν τομείς όπου η πολιτιστική διπλωματία των κρατών μελών είναι η πιο αποτελεσματική από όλους. Όμως, σε ορισμένες περιφέρειες που ίσως είναι πιο απομακρυσμένες, που είναι πιο ευρείες γεωγραφικά, εκεί ίσως μπορεί να βοηθήσει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μπορούμε από κοινού ως Ευρώπη να προωθήσουμε τις δημοκρατικές αξίες και τις ευρωπαϊκές αξίες ως μέρος για παράδειγμα της αναπτυξιακής ε, πολιτικής. Πολλά στοιχεία της εκπαιδευτικής ή της ε, ε, πολιτιστικής πολιτικής μπορούν να ενταχθούν στην αναπτυξιακή πολιτική. Και να μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, τα αθλήματα γεφυρώνουν τα έθνη, γεφυρώνουν τις περιφέρειες, τις περιοχές οι οποίες ιδαλλιώς δεν θα είχαν ευκαιρία να συναντηθούν. Και τέλος να αναφερθώ στη διαδικασία της Μπολόνιας εν συντομία γιατί σας υποσχέθηκα την περασμένη φορά ότι θα σας ενημερώσω σήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνιας. Κάτι το οποίο θα είναι μέγα ζήτημα ενδεχομένως ε, στα, ε, στο όλο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Κριστίνα για την έκθεσή της και τον Έρνεστ Μαραγκάλ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Α, δυστυχώς δεν είναι εδώ. Γιατί στο Γερεβάν ήταν παρόν ε, στην ε, υπουργική διάσκεψη με αντικείμενο τη διαδικασία της Μπολόνιας. Η διαδικασία της Μπολόνιας είναι μια τεράστια επιτυχία κατά τη γνώμη μου γιατί μας δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν οι χώρες να έχουν διάλογο για την ανώτερη εκπαίδευση έτσι ώστε ο χώρος αυτός ο εκπαιδευτικός να γίνει πιο ορατός και να προσεγγίσει το ένα εκπαιδευτικό σύστημα το άλλο σε επίπεδο βάθμιας ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, σίγουρα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση των πεπραγμένων, γιατί τα επίπεδα του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι τόσο διαφορετικά, το ένα δηλαδή σύστημα από το άλλο, ε, που για να προχωρήσει όλη η διαδικασία από κοινού μπροστά πρέπει να σταθούμε μια στιγμή, να κάνουμε αποτίμηση, να βρούμε σωστές λύσεις έτσι ώστε να έχουμε ένα παιχνίδι επίσης όρης, να έχουμε μια τυποποίηση ε, των εκπαιδευτικών συστημάτων. γιατί πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά την ισοτιμία των πτυχίων, των διπλωμάτων και να έχουμε εκπαιδευτικά συστήματα ε, που θα αλληλεπιδρούν περισσότερο μεταξύ τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα είναι περισσότερο συμβατά ε, το και ισότιμα και αντίστοιχα το ένα με το άλλο σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά καταρχάς από μένα και... Να απαντήσω στις εισαγωγικές ερωτήσεις της Προέδρου ως προς τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Βασικά προγράμματα τα βασικά προγράμματα βρίσκονται σε κάπως σταθερή κατάσταση. Έχουμε το Erasmus Plus, το Erasmus Sin και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Όλα αυτά είναι σε σταθερές συνθήκες οικονομικές. Έχουμε καλό προϋπολογισμό για το Erasmus Sin, άρα το μέλλον του προγράμματος αυτού δεν κινδυνεύει και Συνεχώς δίνουμε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση, άρα ε, ε, κάθε δαπάνη που γίνεται στην εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές της οικονομίας και την απασχόληση και την αγορά εργασίας είναι δαπάνη που ε, θα είναι στη διάθεση των κρατών μελών με τα προγράμματά τους και το έργο τους. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, θέλουμε περισσότερους πόρους να δώσουμε στη διαδικασία μετά το Παρίσι. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα προφίλ στα εκπαιδευτικά συστήματα το οποίο θα ενσωματώνει την έννοια της ε, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και θέλουμε να έχουμε αυτό το project, αυτό το έργο για την ηθαγένεια, για τη δημοκρατική κοινωνικοποίηση και για την κοινωνική ένταξη. Και ελπίζω ότι θα έχουμε και προϋπολογισμό για θέματα πολιτισμού. Τώρα για την Ευρώπη 2020 και για το ET 2020. Αυτά εν μέρει ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Τάισεν. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μας και νομίζω ότι είναι ε, αδιέρετα σε κάποιο βαθμό μπορούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας γιατί η επαγγελματική κατάρτιση, η αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα συνδέονται άρρηκτα το ένα με το άλλο. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Γιατί αν ξεχωριστεί η προσέγγιση και η ατομική δεν θα έχουμε επιτυχία. Προστασία της πολιτικής κληρονομιάς. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για το ζήτημα αυτό και εμείς ε, το Συμβούλιο μόλις απάντησε όταν τον προηγούμενο μήνα ε, δημοσιεύθηκε μια ανακοίνωσή μας για την ε, πολιτιστική κληρονομιά. Το Συμβούλιο έχει απαγορεύσει την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών από την Μέση Ανατολή και πριν από μια εβδομάδα όταν βρέθηκα στο Όσλο στην ε, ε, τελετή για το Europa Νόστρα. τόνισα την σημασία και την ανάγκη ενισχυμένης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς υπάρχει όλο και στενότερη συνεργασία μεταξύ της UNESCO και των ε, ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και βεβαίως θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία μας και με τη δική σας επιτροπή στο θέμα αυτό. Το στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων του Juncker ε, βρισκόμαστε σε επαφές με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τα κράτη-μέλη και καλούμε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αιτήσει για το εκπαιδευτικό τμήμα αυτού του σχεδίου επενδύσεων γιατί υπάρχουν πολλές ε, ευκαιρίες όσον αφορά τις μαθητείες στους δημιουργικούς τομείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δυσκολότερο θέμα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η εκπαιδευτική και πολιτιστική υποδομή γιατί ε, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων υποδομών και από τα περιφερειακά ταμεία το στρατηγικό ταμείο, ε, το ταμείο στρατηγικών επενδύσεων δηλαδή θα χρειαστεί να κινητοποιήσει και να απελευθερώσει κονδύλια για, τις, ε, για να γίνουν επενδύσεις ε, στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας και να διατεθούν κονδύλια και χρήματα για την κινητικότητα των μαθητών, των φοιτητών, για την εκπαίδευση των καθηγητών και των δασκάλων και για τις ε, ερευνηστικές ε, διαδικασίες και όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δηλώσει ότι με χαρά θα τα στηρίξει. Και τέλος μια σύντομη παρατήρηση για την συνεργασία μου με τον κύριο Έτιγκερ, τον Επίτροπο Έτιγκερ. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική η πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα αφορά κυρίως το δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την Ιθαγένεια με τις γενικές διευθύνσεις μας. Εγώ ε, είμαι υπεύθυνο για το πολιτιστικό ε, περιεχόμενο στα οπτικοαστικά και για τα πνευματικά δικαιώματα είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον γιατί θα, είναι, ε, θα, έχουμε την, θα αποτελέσει την πρώτη φάση της ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής ε, αγοράς οπότε το θέμα αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και εδώ στο πλαίσιο της δικής σας επιτροπής στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτή την παρουσίαση των πολιτικών σας θεωρώ ότι κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες ε, σίγουρα είναι και δικές μας, διότι και εμείς αυτούς τους μήνες ασχολούμαστε με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αναφερθήκατε στο ψήφισμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, στη Συρία και στο Ιράκ. Πρόκειται ακριβώ για ένα ζήτημα το οποίο είναι μία πτυχή της πολιτιστικής διπλωματίας, ε, την οποία προωθούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου και σίγουρα θα δώσουμε και το λόγο στη συνάδελφο Λιμπάτσκα γιατί για μας ε, η συνέχεια της διαδικασίας της Μπολόνιας είναι υψής της σημασίας διότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, και τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να έχουμε και ένα συγκρίσιμο επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να υπάρχει και μια πραγματική κινητικότητα και ε, προσιτή για τους νέους φοιτητές και σπουδαστές. Επίσης υπάρχει και αυτή η συζήτηση την οποία θα κάνουμε και με μια ακρόαση που θα γίνει τον Σεπτέμβριο για τα 10 χρόνια της σύμβασης της UNESCO για την ε, πολιτιστική και γλωσσική ε, ποικιλομορφία και το πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ε, πολιτιστική ποικιλομορφία μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι από αυτών των θεμάτων θα έχετε και συγκεκριμένε προτάσεις και κατευθύνσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε από τον συναδελφό Σβέρ και την κυρία Λιμπάτσκα μετά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο σας να σας βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο. Εκείνο είναι το μικρόφωνο Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας του και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι μιλάει μια γλώσσα που είναι κατανοητή σε μένα και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει ένας επίτροπος ε, του δικού του διαμετρήματος ε, αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα. Οι προτεραιότητες που μας παρουσίασε είναι ορθές. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για μεγαλύτερη αποσχόληση. Επομένως είναι ο ρόλος των σχολείων να εκπαιδεύουν ανθρώπους όχι μόνο για το χώρο εργασίας αλλά και για τη ζωή. Συμφωνώ επίσης και με τη δημοκρατική κοινωνικοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο μα το παρουσίασε, ε, αυτό το οποίο συμβαίνει στους νέους αυτή τη στιγμή εν καιρό κρίσης είναι μια αποξένωση. αποξένωση. Γίνονται παθητικοί, είναι αποκλεισμένοι και δεν εντάσσονται στην κοινωνία, δεν αφομοιώνονται στο δημόσιο βίο. Και φυσικά αυτό ε, από μόνο το αποτελεί καταστροφή. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση από πλευρά των νέων και στην πολιτική. Το σχολείο είναι ε, ο χώρος αριστείας της κοινωνικοποίησης και εμείς ε, είμαστε οι πλέον αρμόδιοι προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς και το σχολείο δεν είναι ο μόνος ε, ένοχος και ο μόνος υπεύθυνος ε, για τον αποκλεισμό των νέων. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οικογενειακός ε, κύκλος, αλλά η παιδεία είναι αυτή η οποία πραγματικά θα μπορέσει να βοηθήσει και να συνδράμει προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης διότι άκουσα ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους Ευρώπη 2020. Βεβαίως οι στόχοι αυτοί δεν είναι και ιδιαίτερα απαιτητικοί. Ίσως ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε στη διάρκεια αυτής της θητείας ε, και ένα νέο ορισμό αυτών των στόχων. Παραδείγματος χάρη, ο δείκτης ε, των νέων που πηγαίνουν σε ανώτατη παιδεία αυτό από μόνο του δεν αρκεί ως δείκτης. Ε, ε, κάποιος πρωθυπουργός είπε προσφάτως ότι το 80% δηλαδή η πλειονότητα των νέων ε, προχωρούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δεν αναφερόμαστε στην πραγματικότητα, στην ποιότητα αυτής της εκπαίδευσης. Ε, μπορεί επίσης να πρόκειται για νέους οι οποίοι δεν βρίσκουν μια θέση απασχόλησης και απλώς γράφονται στο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει από μόνο το δείκτης ε, ε, κάτι συγκεκριμένο. Όπως ε, το ίδιο ισχύει και με το δείκτη αυτό της μείωσης των ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο. Από μόνος του δεν είναι ενδεικτικός για τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ένα δείκτη αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ένα δείκτη δηλαδή ο οποίος θα βασίζεται στο περιεχόμενο και που θα προσμετρά πραγματικά την ποιότητα της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τη δική σας την άποψη για το κατά πόσον υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε ένα νέο καθορισμό των στόχων και των δικτών ε, της εκπαίδευσης, διότι ιδίως όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, δεν νομίζω ότι έχουμε ουσιαστικές βελτιώσεις. Παρακαλώ κυρία Λεμπάτσκα. Ah, uh, Today they are lazy. Εκο, <laughs> it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Christine. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι μεγάλη μας τιμή και με μεγάλη χαρά ακούσαμε αυτά που είπατε. Τρεις παρατηρήσεις θέλω όμως να κάνω. Πρώτον, συμφωνώ ότι η διαδικασία της Μπολόνια ήταν εξαιρετικά σημαντική. Αποτελεί το θεμέλιο για την οικοδόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Υπάρχει μια γενική πεποίθηση στην Ευρώπη ότι η, πληροφορία της, ε, η κοινωνία της πληροφορίας βαίνει προς το τέλος της και πλέον το σημαντικότερο ζήτημα είναι ο πολιτισμός της γνώσης. Νικητές θα είναι εκείνοι που θα έχουν θέσει τα πράγματα στη σωστή του βάση όσον αφορά τι γνώσει του. Η διαδικασία τη Μπολόνια λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικά και νομίζω ότι αναδείξατε κι εσεί τη συγκρισιμότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων ω βασικά στοιχεία αυτή τη διαδικασία, Αλλά για να υλοποιηθούν στην πράξη όλα αυτά απαιτεί απαιτείται μεγαλύτερη δημιουργικότητα όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων αυτών και θα πρέπει να υπάρξουν και μηχανισμοί παρακολούθησης της κινητικότητας των φοιτητών και των μαθητών. Θα πρέπει δηλαδή με άλλα λόγια να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στους φοιτητές που έχουν ε, παρακολουθήσει μαθήματα σε διάφορα ιδρύματα και αν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους κατάφεραν να βγουν στην αγορά εργασία και αν τελικά ε, τα μαθήματα που παρακολούθησαν, οι κύκλοι σπουδών που παρακολούθησαν ήταν συγκρίσιμοι. Ένα άλλο ζήτημα που, ε, που αναφέρατε ήταν ότι θα πρέπει να... Ε, ότι η απασχόληση υπάγεται πάντοτε στην, εργασία, στην πολιτική για την απασχόληση. Πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ε, δημοφιλία της ε, διτής εκπαίδευσης θεωρητικής και πρακτικής μαζί και εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει ε, η διτή εκπαίδευση αυτή να προσφέρεται σε όλους τους ε, τομείς της εκπαίδευσης. Αλλιώς ε, θα, οι ανθρωπιστικές σπουδές θα μείνουν πίσω και αυτό είναι κάτι που δεν, δεν, δεν το επιθυμούμε κανείς μας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αναφερθήκατε ε, στην διαδικασία του Παρισιού ως μια εξαιρετική διαδικασία. Αυτά τα 21 σημεία που ε, προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή. Έχετε συζητήσει με τους συναρμόδιους επιτρόπους πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο αυτό ή το ε, ίντερνετ για την για το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Ήπειρό μας μια διαφορετική αφήγηση από αυτή που προτείνουν οι τζιχαντιστές. Δυστυχώς, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι ε, περνούν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ε, μια πλατφόρμα ώστε να τους... Ε, ώστε να τους ε, προσελκύσουμε εμείς και να τους αποσπάσουμε από την επιρροή των, εξτρε, ε, εξτρεμιστών. Άρα τα ερωτήματά μας είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία της Μπολόνια και πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το δίκτυο για την ενίσχυση της δημοκρατίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Ευχαριστώ κύριος Λούερ. Is Yes, good. Okay. Um, Καλώς ήρθατε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Η κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι μια έννοια που εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου την αμφισβητούν. Ιδιαίτερα ε, αυτές τις φεντεραλιστικές ε, απόψεις ε, και τα όσα μας είπε και ο Έλληνας συνάδελφός σας, ο κ. Αβραμόπουλος χθες. Υπάρχει ε, μία ε, κίνηση ε, αντίθετη προς ένα μοντέλο 28 κρατών μελών που θα συνεργάζονται ελεύθερα και είτε αρέσει σε κάποιους εδώ μέσα είτε όχι, αυτό συμβαίνει ήδη. Η ισχυρές εθνικές πολιτικές ταυτότητες ε, δεν, χωρίς να είναι κλειστές μπορούν να συνεργαστούν και μπορούν να συνδράμουν και στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού. Και για να εξετάσουμε με πιο πρακτικούς όρους αυτό το συνεργατικό μοντέλο και για να δώσουμε μια πιο απτή προσέγγιση ε, ε, των εκπαιδευτικών συστημάτων Αναφερθήκατε στην Πολόνια, το οποίο εμείς ε, ως ECR συ, ε, υποστηρίζουμε ε, θερμότατα. Αν δει κανεί όμως τις περικοπές που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, φαίνεται ότι πολλά από τα κονδύλια που προβλέπονται απευθύνονται κυρίως σε συγκεκριμένες χώρες μέλη, σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδίως σε εκείνα που ε, έχουν μια έντονη κρατική παρουσία στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Πώς λοιπόν εσείς σκοπεύετε να προχωρήσετε σε διάλογο με τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με τους υπουργούς παιδείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσετε να ενισχύσετε και την ε, πρόσβαση στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ναυράτσης για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας ε, θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι μάλλον περισσότερο ερώτηση και άλλη μια σκέψη, ε, την οποία δεν ξέρω αν θα συμμεριστεί και ο Επίτροπος. Να περάσω καταρχάς στην ερώτηση. Αναφερθήκατε στη σημασία της πολιτιστικής διάστασης της εξωτερικής ε, δράσης και της πολιτιστικής διπλωματίας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς ε, είπα της εκπροσώπου της κυρίας Μογκερίνη. Θα ήθελα να εμβαθύνετε λίγο περισσότερο στην έννοια της ε, πολιτιστικής δημοκρατίας. Πώς βλέπετε εσείς ε, τη συγκεκριμένη αυτή άνοια, λίγο πιο συγκεκριμένα, και τι ρόλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να διαδραματίσει ο πολιτισμός στη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ε, ιδίως ε, σε τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η μετανάστευση και η κινητικότητα των ατόμων. Και επίσης ε, βρήκα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πρώτα πράγματα που μας είπατε για την ανακεφαλαίωση που κάνατε για μια σειρά από ε, τραγικά γεγονότα για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σας. Αναφερθήκατε στην περίπτωση του Παρισιού, της Κοπενχάγης, την περίπτωση των Βρυξελών το σκεπτικό σας ήταν ότι θεωρείτε ότι υπάρχει μία απόσταση ε, σε σχέση με τις ε, ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Συμφωνώ βέβαια με αυτό το οποίο είπατε, αλλά ίσως θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτό τον κατάλογο που αναφέρατε εσείς και κάποια ζητήματα τα οποία δεν θεωρώ ότι συντονίζονται υπερβολικά με τις ευρωπαϊκές αρχές κατά την απόψή μου. Παραδείγματος χάρη η διαβούλευση για την θανατική ποινή, η πιθανή ε, ε, επαναφορά της θανατικής ποινή σε κάποιες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης η μετανάστευση, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον προηγούμενο μήνα και ε, υπήρξε μια αναφορά στη χώρα καταγωγής σας, ε, στην Ουγγαρία, και μάλιστα και συγκεκριμένη αναφορά στην κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχατε κι εσείς πριν γίνετε επίτροπος. Αυτές οι δύο διαβουλεύσεις, αυτές οι δύο έρευνες που έχουν ξεκινήσει στην Ουγγαρία έχουν καμία σχέση με τις δημοκρατικές ε, αρχές ε, που ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκλέζος. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα την εισήγηση. Αφορούσε τον τομέα μονάχα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν έκανε όμως καθόλου δεν άγγιξε το θέμα του τομέα δημιουργίας πολιτισμού. Δηλαδή, εάν ασχοληθούμε μονάχα με την πολιτιστική μας κληρονομιά και δεν σκεφτούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτισμό, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Ένας λαός που στηρίζεται μονάχα στην κληρονομιά του είναι ένας λαός προγονόπληκτος. Πάσχει από προγονοπληξία και δεν έχει καθόλου μπροστά του μέλλον. Δεν είπατε ούτε μια κουβέντα για τη διατήρηση, τη διατήρηση είπατε, για την δημιουργία πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα σταθώ πρώτα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχω ξανατονίσει σε αυτήν την Επιτροπή και ξανατονίζω και πάλι ότι πρώτη δουλειά είναι τα έργα που έχουν δημιουργηθεί τα έργα τέχνης πρέπει να γυρίσουν στον τόπο παραγωγής τους, καταγωγής τους, εκεί που δημιουργήθηκαν. Αυτό σημαίνει όχι μονάχα η επιστροφή των κλεμμένων αρχαιοτήτων, των ληστευμένων αρχαιοτήτων από τις γερμανικές στρατιές κατοχής από το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα, αλλά σημαίνει και επιστροφή Μιλάω για την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και για όλες τις χώρες. Ε, και την επιστροφή και της Αφροδίτης της Μήλου και της, αμο, ε, Σαμοθράκης και των αετομάτων του Παρθενώνα. Αυτό είναι το ένα θέμα που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Όσον αφορά την, τον τομέα πολιτιστική δημιουργία, θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι πολιτισμό καινούριο δημιουργούν μονάχα οι πολίτες μιας πόλης όταν ασκούν οι ίδιοι πολιτικοί και δεν την αφήνουν την άσκηση πολιτικής σε επαγγελματίες πολιτικούς. Τότε δημιουργείται πολιτισμός. Συνεπώς, στον τομέα ειδικά το δικό σας της παιδείας, αν δεν σταματήσει η παπαγαλία δεν πρόκειται ποτέ οι φοιτητέ που θα εξέρχονται, οι μαθητές που θα εξέρχονται να είναι δημιουργοί. Οι παπαγάλοι δεν δημιουργούν, μιμούνται οι παπαγάλοι. Μόνο μίμηση κάνουν οι παπαγάλοι, δεν δημιουργούν. Η κατάργηση λοιπόν της παπαγαλίας και η αντικατάστασή της με εργασία των μαθητών και των φοιτητών είναι η μόνη λύση και για να καταργήσει και την παραπαιδεία. Και επίσης η ελεύθερη δυνατότητα για κάθε οργανισμό που θέλει να φτιάξει παιδεία. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε κάτω από Οθωμανική κυριαρχία και όμως δημιουργήσαμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στη Μικρά Ασία παρά τη βούληση και τη θέληση του κατακτητή. Επίσης η διατήρηση των συνθήκων δημιουργίας του πολιτισμού. Αναφέρω εδώ τη Μελίνα τη Μερκούρη την οποία γνωρίζετε πιστεύω όλοι η οποία πρωτοστατούσε στα θέματα της πολιτιστικής πρωτεύουσα για να πω δεν χρειάζεται μονάχα η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι κάτι που είχε συμφωνήσει επίσης η Μελίνα χρειάζεται και κάθε, σε κάθε περιφέρεια να, να δημιουργήσουμε μια πόλη πολιτισμού αλλά και σε κάθε χωριό. Επιμένω, σε κάθε χωριό. Όχι μονάχα σε ένα χωριό της Ευρώπης, σε κάθε κράτος της Ευρώπης ένα χωριό. Και συγκεκριμένα θα έλεγα και δεν το κρύβω το χωριό μου έχει δημιουργήσει πέντε μουσεία και έχει υποκατασκευή άλλα τρία με 1200 κατοίκους. Το κατανοείτε αυτό, πέντε μουσεία και άλλα τρία υποκατασκευή. Κανονικά θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να δει τον τόπο και να κατασκευάσει αν είναι δυνατόν και τα κτίρια για να στεγαστούν τα μουσεία αυτά τα οποία στεγάζονται δόθε κήθε. Η πρότασή μου συγκεκριμένη. Όλη μας η Επιτροπή, σας το έχω ξαναπεί, να έρθει να επισκεφθεί το χωριό, να επισκεφθεί το χωριό σας προσκαλώ τα έξοδα δικά σας έως την άξο, από εκεί και πέρα δικά μου τα έξοδα, ναι. δηλαδή του το χωριό θα σας αναλάβει και να δείτε τον τόπο και ειδικά για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τα έξοδα, να κτίσει τα κτίρια αυτά. Είναι μια πρόκληση στην οποία να απευθύνω και θα επανέρχομαι συνεχώς. Θα με υποστείτε ακόμα ένα μήνα. Έχω υποβάλει σήμερα την παρέτησή μου, σε ένα μήνα παρετούμε, όπως είχα δηλώσει από παλιά η διάρκεια της θητείας μου είναι γιατί για μένα η θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι επάγγελμα. Χρειάζεται να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας, μήνα, ένας χρόνος μου αρκεί. Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα δηλαδή παρετούμε, θα με υποστείτε ακόμα ένα μήνα. Να το έχετε υπόψη θα με υποστείτε ένα μήνα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Καρό Γκλέζος. Αγαπητέ κύριε Γκλέζο, εμείς δεν χρειάζεται να σας υποστούμε. Αποτελεί τιμή για μας ε, να σας έχουμε εδώ και χαιρόμαστε που έχετε επιλέξει την Επιτροπή Πολιτισμού για να εκφράσετε τις απόψεις και τις θέσεις σας. Η Νάξος ε, είναι διαβόητη σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να είναι ένα μικρό νησί, αλλά είναι ένα παγκόσμιο νησί. Ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε τώρα σήμερα και χαίρομαι και λυπάμαι πολύ συγγνώμη που θα μας εγκαταλείψετε. Ε, Βέβαια είπατε ότι θέλετε να δώσετε και τα ενία σε κάποιον άλλο συνάδελφο και αυτό είναι μεγάλο ψυχή από πλευρά σα. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την κυρία Τρούπελ και μετά θα συνεχίσουμε με τι υπόλοιπε παρεμβάσει. Τώρα θα κλείσω αυτό ο γύρος με την κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω για το θέμα των μαθητών και τον κίνδυνο αποξένωσής τους από την κοινωνία ή και στρατολόγησή τους από εξτρεμιστές και την ε, ε, ελκυστικότητα που ε, τους ασκούν οι ιδεολογικές, οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες και χρειαζόμαστε συνεργασία με τη μουσουλμανική κοινότητα γιατί πολλές φορές επηρεάζουν τους νέους ανθρώπους, ε, τους καθοδηγούν και τους υποστηρίζουν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες όπου ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές για την ίδια τους τη θρησκεία, διότι όταν οι μουσουλμάνοι μαθητές γνωρίζουν πράγματα για την ίδια τους την ε, θρησκεία δεν εντυπωσιάζονται τόσο πολύ από τους αλαφιστές. Και μια ερώτηση. Αντιμετωπίζουμε σε διάφορα κράτη-μέλη πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα για το πρόγραμμα ε, Erasmus ότι δεν συμπεριλαμβάνονται μικρά ε, project, μικρά προγράμματα και ότι υπάρχει σαφή στάση να χρηματοδοτούνται τα μεγάλα έργα. Ε, μικρά ιδρύματα ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα και νομίζω ότι θα πρέπει κι εσείς ξεκάθαρα να πείτε ότι δεν, πρέπει να ανακοπεί αυτή η τάση, χρειάζεται αλλαγή σε αυτόν τον ε, τομέα και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε επ' αυτού. Και τελευταία παρατήρηση αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος πνευματικών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί είπατε ότι τον επόμενο μήνα, τους επόμενους μήνες θα εκφραστείτε ως Κομισιόν επί του θέματος αυτού, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η αρχή της εδαφικότητας. Από την άλλη πλευρά θέλουμε να δημιουργήσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και ε, από μια άποψη βεβαίως υπάρχει μια αντίφαση. Από την άλλη πλευρά για να διατηρηθεί η πολιτιστική πυκλομορφία και το περιεχόμενο από μικρές περιοχές, φυσικά χρειαζόμαστε αυτή την αρχή της ε, εδαφικότητας. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας άποψη αυτή τη στιγμή για αυτό το πολύ λεπτό ερώτημα, για αυτή την ισορροπία μεταξύ των δύο αρχών. Επίτροπε, να σας δώσω τώρα το λόγο γιατί υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να δώσω σύντομες συγκεκριμένε απαντήσεις για να υπάρξει χρόνος για περισσότερες ερωτήσεις στη συνέχεια. Ετέθησαν δύο ερωτήσεις για την ε, ταξινόμηση των ε, πανεπιστημίων και πιθανή αναδιάρθρωση αυτής της ταξινόμησης. Υπάρχει μια, ένας κατάλογος με μια αμερικανική βαθμολόγηση και υπάρχει και το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Ακόμα και μεθοδολογικά θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ευρωπαϊκές μεθόδους ε, διδασκαλίας και ανώτατης εκπαίδευσης από τις Αμερικανικές, διότι, για παράδειγμα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της κατάταξης των ε, Αμερικανικών ε, συστημάτων είναι οι δημοσιεύσεις ε, και η βιβλιογραφία, ενώ οι σχέσεις με τους φοιτητές και η κοινωνία της γνώσης και οι ανταλλαγές απόψεων μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών δεν βαθμολογείται στην Αμερικανική κατάταξη. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά διακριτικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν είναι απλώς μεταφορά γνώσης, αλλά είναι μια κοινότητα μεταξύ ε, σπουδαστών, ε, φοιτητών και ακαδημαϊκών. Υπάρχει μια συνεχή συζήτηση επί του ζητήματο και είμαστε καθόλου ανοιχτοί. Αν μπορέσουμε να το καθορίσουμε από μεθοδολογική σκοπιά και μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποθέσεις για την ε, κατάταξη, νομίζω ότι θα έχουμε κάτι θετικό. Θα έχουμε μια πιο ήπια, μια πιο ευρωπαϊκή ε, κατάταξη που θα είναι πιο ευαίσθητη στα ευρωπαϊκά διακριτικά χαρακτηριστικά. Τώρα, τα διτά συστήματα και ε, το κατά πόσον μπορεί να γίνουν πιο δημοφιλή. Νομίζω ότι τα διτά συστήματα αυτή τη στιγμή ε, είναι μάλλον τα πιο δημοφιλή συστήματα στην Ευρώπη, διότι ε, έχω συναντήσεις με υπουργούς παιδείας και απασχόλησης που έχουν εισαγάγει αυτά τα διτά συστήματα και έχω και συναντήσεις με υπουργούς εκπαίδευσης και ε, παιδείας και απασχόλησης που σκέφτονται την εισαγωγή αυτών των διτών συστημάτων. Ε, γνωρίζω για παράδειγμα ότι για την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία υπάρχουν ε, ε κάποιες ε, προβληματικές πτυχές αυτών των διτών συστημάτων. Θα πρέπει να κάνουμε και μια αξιολόγηση των διτών συστημάτων. Το εκπαιδευτικό σκέλος είναι αρκετά σαφές ε, στο διτό σύστημα. Το ε, θέμα της μαθητείας όμως και της πρακτικής άσκησης είναι απόλυτα εξαρτημένο από τη συνεισφορά των επιχειρήσεων και του βιομηχανικού κλάδου, τις ε, διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται μιας μορφής τυποποίηση του διτού συστήματος ή τουλάχιστον κάποια κοινά σημεία αναφοράς. Η διαδικασία μετά το Παρίσι και το διαδίκτυο. Μόλις εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, το οποίο αφορά και βράχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες προκλήσεις της ασφάλειας ε, στην Ευρώπη και υπάρχουν πάρα πολλά μέσα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα εξτρεμιστικά φαινόματα. Η ε, παιδεία είναι η πιο μακροπρόθεσμη βέβαια γιατί οι συνέπειες ε, θα φανούν ε, μακροπρόθεσμα αλλά επί παραδείγματι προστασία προσωπικών δεδομένων, το διαδικτυακό έγκλημα, η επιβολή του νόμου, για τα θέματα αυτά είναι βραχυπρόθεσμα καθήκοντα και εξ όσων γνωρίζω η Επίτροπος Γιούροβα προχωρά τις συζητήσεις για την προστασία των δεδομένων και την ε, διαδικτική προστασία των ε, καταναλωτές, κάτι το οποίο φυσικά θα μπορέσει να βοηθήσει και την προστασία των νέων ανθρώπων στο διαδίκτυο. Κύριε Λιούερ, για μένα η κοινή πολιτιστική κληρονομιά και ο φεδεραλισμός είναι συνώνυμα. Παραδείγματο χάρη, ο Φραν Λίστ ή ο Λίστ Φέρεντ, όπω είναι γνωστό στην Ουγγαρία, πρόκειται για μία ένα συζήτηση μεταξύ Αυστριακών και Ούγγρων. Αν ο Φραν Λίστ ή ο Λίστ Φέρεντ ήταν Αυστριακό ή Ούγγρο συνθέτη. Εγώ πρέπει να σα πω ότι είναι Ευρωπαίο συνθέτη, διότι η προσωπική του συνεισφορά είναι συνεισφορά προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όχι μόνο στον αυστριακό ή τον ουγγρικό πολιτισμό, αλλά προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Αυτό ε, δεν σημαίνει φεντεραλισμός. Εγώ θα έλεγα ότι η θέση μου δεν είναι ομοσπονδιακή. Εγώ θεωρώ ότι προωθώ κάποια πράγματα. Είμαι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των Υπουργών Παιδείας και ε, Πολιτισμού και εσείς είστε οι διαμεσολαβητές μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, διότι γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η επικουρικότητα και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά είναι μια σύνθεση των εθνικών και περιφερειακών πολιτιστικών κληρονομιών και φυσικά δεν είναι ένα ομοιογενές μείγμα, είναι ε, ένα αμάλγαμα πολύ διαφορετικών αλληλένδετων όμως ε, πολιτιστικών ε, στοιχείων κληρονομιάς και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικό. Όσον αφορά το σχέδιο επενδύσεων Juncker, Είμαστε σε επαφή με πανεπιστήμια και κυβερνήσεις των κρατών μελών και αυτή τη στιγμή οργανώνουμε ένα εργαστήριο το οποίο θα γίνει το φθινόπωρο, κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο εδώ στις Βρυξέλλες και σκοπεύουμε να διοργανώσουμε περισσότερα εργαστήρια περιφερειακά για την Κεντρική Ευρώπη, για τη Βόρεια Ευρώπη, για την ε, Δυτική Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη, ώστε να προωθήσουμε την ιδέα των επενδύσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, διότι υπάρχουν ε, ε, διάφορα μοντέλα, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε καλές λύσεις και γι' αυτό και με τους ε, κατάλληλους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κύριε Μάουρα, νομίζω ότι η πολιτιστική διπλωματία και η πολιτική γειτονίας, η αναπτυξιακή πολιτική, και οι πολιτιστικές ε, δραστηριότητες και διπλωματία μπορούν να συνεπάρξουν και μάλιστα πολύ ειρηνικά. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής εξέλιξης είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και αφενός ε, μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει πιο δημοφιλής ε, αν ενταχθεί στα πλαίσια της πολιτιστικής διπλωματίας και αφετέρου μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό μέσο για να προσεγγίσουμε άλλες περιοχές, άλλες ε, ε, περιφέρειες, άλλους λαούς. Και η πολιτιστική κληρονομιά αφορά την τέχνη, τον πολιτισμό, την ειρηνική συνύπαρξη, την ύπαρξη ε, καλών και θετικών αξιών της ανθρωπότητας. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό θέσατε και μία ερώτηση για τις ουγγρικές εξελίξεις. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, διότι σας υποσχέθηκα στη διάρκεια της ακρόασής μου ότι θα είμαι απόλυτα ανεξάρτητος για τη χώρα μου, όσον αφορά τη χώρα μου και την κυβέρνησή μου και επομένως αυτό σημαίνει ότι δεν σχολιάζω ε, και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία, στη Σουηδία. Αντίστοιχα λοιπόν δεν σχολιάζω και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία. Εάν υπάρχουν εκπαιδευτικά πολιτιστικά ζητήματα στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, Βεβαίως και με στη διάθεσή σας για να βοηθήσω να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, ε, όλα τα κράτη-μέλη ε, έχουν θέματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, δημοκρατικής κοινωνικοποίησης στα σχολεία, αλλά η θανατική ποινή και η μετανάστευση δεν αποτελεί θέμα του χαρτοφυλακίου μου, λυπάμαι πολύ. Κύριε Γλέζο Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την τεράστια συνεισφορά του ελληνικού πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό αποτελεί θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα από τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ακριβώς ε, για λόγους επικουρικότητας δεν ε, θα ήθελα να παρέμβω σε διακυβερνητικά ζητήματα όσον αφορά την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς ή την ανταλλαγή ε, πολιτιστικών αντικειμένων, έργων τέχνης και ούτω καθεξής εάν υπάρχει κάποια συζήτηση μεταξύ κρατών μελών ως προς το πού θα πρέπει να βρίσκονται διάφορα πολιτιστικά έργα τα οποία προστατεύονται μέσω νομοθεσίας και διεθνών προδιαγραφών, οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να κάνουν το διάλογο μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ε, κατασκευή μουσείων. στα περιφερειακά ταμεία, στα ταμεία συνοχής υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Και είμαι βέβαιος ότι εάν υπάρχει ανακαίνιση ή ε, κατασκευή νέων κτηρίων ε, στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, ε, διότι υπάρχει και μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για τις μικρής κλίμακας πολιτιστική επενδύσεις, που σημαίνει ότι τα περιφερειακά ταμεία υποστηρίζουν στις ε, χώρες που δεν ε, έχουν υπερβεί το όριο των 5 εκατομμυρίων. Υπάρχει μια συζήτηση εν εξελίξει αυτή τη στιγμή και τα υποστηρίζουμε αυτά. Κύριε Τρούπελ, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν πάρα πολύ καλά παραδείγματα από τις ε, σκανδιναβικές χώρες για διαθρησκευτικές γνώσεις, διαπολιτισμικές γνώσεις ε, στο πρόγραμμα σπουδών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ε, διότι περισσότερες γνώσεις μπορούν να φέρουν και ε, καλύτερα αποτελέσματα. Αν γνωρίζουμε το πραγματικό Ισλάμ, αν γνωρίζουμε την πολιτιστική διάσταση του Ισλάμ, σίγουρα θα μπορέσουμε ε, να ε, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες και ισχυρίζονται οι τζιχαντιστές. Ε, είχα κάποιες επαφές για τη διαδικασία μετά το Παρίσι και οι εκπρόσωποι των νέων ε, μουσουλμάνων ήταν εκεί. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη συνεισφορά των, ε, της μουσουλμανικής κουλτούρας σε αυτό τον διάλογο μεταξύ θρησκειών. Όσον αφορά τα μικρότερα προγράμματα και τα ε, διάφορα προγράμματα, νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα στη διάρκεια της επίσκεψής σας ε, θα διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα από τα φλέγοντα ζητήματα σήμερα το απόγευμα, τη συνεισφορά μας και το τι ακριβώς μπορεί να κάνει το Erasmus Plus. Copyright τώρα, πνευματικά δικαιώματα. Νομίζω ότι θα ήταν σφάλμα να υποστηρίζουμε μια μέθοδο ε, πανάκια για τον όλο τομέα του πολιτισμού. Διότι είναι τόσο προηγμένα τα συστήματα πνευματικών δικαιωμάτων και υπάρχουν ε, ε, διαφορές από κλάδο σε κλάδο. Υπάρχουν ε, θέματα για την ε, μουσική βιομηχανία, για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, ε, για τα βιβλία και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της πρόσβασης των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των δημιουργών μια κατάλληλη ισορροπία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την δέουσα ισορροπία Κατά την άποψή μου ένα στοιχείο είναι η φορητότητα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να λύσει ίσως το, το δίλημα της εδαφικότητας σε σχέση με την νέα αγορά, διότι αν κάποιος θέλει να αγοράσει πολιτιστικό περιεχόμενο ε, μπορεί να το λάβει από μόνος του και το άλλο στοιχείο ε, νομίζω ότι είναι ο εξυγχρονισμός χωρίς να υπάρξει όμως διαγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεχρονίσουμε τα συστήματα προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, διότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή και υπάρχουν πάρα πολλέ εξελίξει, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να προστατευτούν ε, οι βασικοί θεσμοί και τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας ε, του συστήματο του copyright. Ευχαριστώ πολύ για αυτέ τι απαντήσει, στι ερωτήσει μα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στου υπόλοιπου συναδέλφου. Έχουμε άλλα πέντε άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η κυρία Καμερέβερ το όχι. Δίνει το καλό παράδειγμα και δεν θα μιλήσει. Η συνάδελφος Εύανς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε για την παρουσίασή σας. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα όσα συμβαίνουν μετά τη διαδικασία του Παρισιού. Είναι ένα ζήτημα που συζητούμε όλοι σε όλες τις χώρες. Προκαλεί μεγάλες ανησυχίες και είναι σημαντικό να ανταλλάσσουμε εμπειρίες όσον αφορά την ε, εκπαίδευση και την, αποκαλ, τον την αποκαλούμενη ριζοσπαστικοποίηση. Και άκουσα να λέτε ότι συνεργάζεται με όλους τους υπουργούς παιδείας γιατί για παράδειγμα στην ε, Ουαλία η εκπαίδευση ε, υπάρχει μια ε, αυτονομία της δικής μας περιφέρειας ως προς το, τα εκπαιδευτικά συστήματα είμαστε και δίχλωση χώρα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συνεργάζεστε άμεσα με τους περιφερειακούς υπουργούς παιδείας αν εμπλέκονται ε, ενεργά στην όλη διαδικασία. Όσον αφορά το ζήτημα των μειωνοτικών γλωσσών, σας ρώτησα το φθινόπωρο τι προβλέπετε να κάνετε όσον αφορά την γλωσσική στρατηγική όχι μόνο για τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αλλά και για τις ε, μειονοτικές γλώσσες, για τις μικρές γλώσσες και ε, είπατε ότι θα δημιουργήσετε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφάλιζε τη μη διάκριση στη βάση ε, της γλώσσας. Αλλά στον οπτικοακουστικό τομέα υπάρχει ένα σύστημα βαθμολόγησης και φαίνεται ότι οι μειονοτικές γλώσσες ε, έχουν ε, χαμηλότερη βαθμολογία από τις επίσημες γλώσσες. Όχι μόνο στην Ουαλία αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει μια κατάσταση όπου οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ε, γιατί δεν δημιουργούν παραγωγές στις μειονοτικές γλώσσες αλλά και οι πολύγλωσσες παραγωγές ε, υποφέρουν. Θα ήθελα να μου πείτε αν, υπάρχουν, λοιπόν, αν υπάρχει καθόλου πρόοδος όσον αφορά τη γλωσσική στρατηγική για την προώθηση των ε, μικρών, των μειονοτικών γλωσσών ε, σε σχέση με τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η Τζούλη Okay, sorry. Συγγνώμη. Λειτουργεί το μικρόφωνο μου ευτυχώς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που μπορώ να πάρω το λόγο γιατί θέλω να πω κάτι για την ταυτότητα. Για την... τις εθνικές μας ταυτότητες και την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους ε, βουλευτές ότι ο πολιτισμός εξελίσσεται διαρκώς. Δεν είναι ένα μέγεθος στατικό. Και όποιος το πιστεύει αυτό, αυτά πατάτε, διότι εμείς είμαστε το αποτέλεσμα όλων όσων προηγήθηκαν ιστορικά, όλων των προκλήσεων που αντιμετώπισαν άνθρωποι σε όλες τις σφαίρες της ζωής και προσωπικά ε, ε, εμένα ε, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η πολλαπλότητα των ταυτοτήτων που έχουμε. Εγώ είμαι και από τη Βόρεια Αγγλία και από την Αγγλία και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την, Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη και είμαι και πολίτης του κόσμου. Είναι υπερβολικά απλουστευτικό να επικεντρωνόμαστε ε, σε έναν φόβο για τις εθνικές ταυτότητες όταν ζούμε σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τόση ποικιλομορφία. Είπατε ότι δεν θέλετε να ε, εκφραστείτε για ζητήματα μεταναστευτικά ή ζητήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένη χώρα, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και οι μετανάστες έχουν διαμορφώσει, συνδιαμορφώσει τον ε, πολιτισμό μας. Και μιας και μιλούμε για τις τέχνες και για τον πολιτισμό, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ζήτημα της ε, μετανέστασης. Ένας από τους συγγενείς μου ήταν μετανάστης που ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλεια... Βασίλειο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και αυτό ε, είναι ένα γεγονός ιστορικό που συνδιαμόρφωσε, που καθόρισε και τον πολιτισμό του Νότιγχαμ, διότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ένιωθαν ασφαλείς πλέον στην ε, χώρα καταγωγής τους. Θα ήθελα να πω ότι οι μετανάστες που υποφέρουν αυτή τη στιγμή χρειάζονται την υποστήριξή μας αναμφίβολα και εκείνοι με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην εξέλιξη της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Είναι και αυτό μια πτυχή της συζήτησης που πρέπει να κάνουμε. Και μιας και ε, είμαι βουλευτής εδώ και ένα χρόνο, ε, θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι το πεδίο της μάχης ε, πολλές φορές ε, πολλοί άνθρωποι μπορεί να ισχυρίζονται ότι ο πολιτισμός ε, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί επικεντρωνόμαστε εδώ στην νομοθεσία αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο πολιτισμός είναι το πιο φλέγον ζήτημα είναι το ζήτημα το οποίο ανησυχεί τους περισσότερους ανθρώπους στο μέγιστο βαθμό ο εξτρεμισμός είναι κάτι που μας ανησυχεί όλους διότι λόγω και των, των, των συγκρούσεων, λόγω των απολειών ε, των θανάτων, λόγω των βασανιστήριων, λόγω της καταπίεσης. Ε, είναι ένα ζήτημα που συζητείται στη δημόσια σφαίρα, στα μέσα μαζικής, ένωσης, ε, μαζικής ενωμέρωσης και είναι και ένα ζήτημα που αφορά και τους νέους ανθρώπους μας. Οπότε θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω πώς εμείς, εμείς και εσείς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων όσον αφορά τη συμμετοχή συμμετοχή τους στο διαπολιτισμικό διάλογο, στις κοινωνίες τους, μεταξύ διαφόρων λαών, μεταξύ διαφόρων ομάδων κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τον διάλογο και με χώρες που ε, αντιμετωπίζουν το, το φάσμα της αστάθειας. Πώς μπορεί να ενισχυθεί το ζήτημα της ατυπικής εκπαίδευσης, της διαβίου εκπαίδευσης για να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι τέχνες είναι το σημαντικότερο εργαλείο, το σημαντικότερο μέτρο, μέσο που έχουμε ε, στα χέρια μας για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Υποστηρίζω από αυτή την άποψη ε, ιδιαίτερος αυτό που είπατε για, την, ε, ε, για τον συνδυασμό της πολιτιστικής και της εξωτερικής πολιτικής και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διευρυνθεί ως στόχος και στους, στην Κομισιόν ευρύτερα. Ο κύριος Μόργαν, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, δεν θα σταθώ σε κάποια πράγματα. Θα κάνω μια πρώτη ερώτηση που είναι προς αντίστοιχη κατεύθυνση μάλλον από αυτό που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Όσον αφορά το σχέδιο Γιούγκερ, για να συνεχίσω με την παρουσίαση της Προέδρου μα ε, σχετικά με τη δυσκολία και το γεγονός ότι τα θέματα της παιδείας και του πολιτισμού δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο πρόγραμμα και χρειάστηκε να διανυθεί κάποιος δρόμος για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων όμως. Έχετε εσείς μια εικόνα του τι ακριβώς ε, θα μπορούσε να θεωρηθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις σε αυτό το σχέδιο Υπάρχει και όλη η συζήτηση για τη στρατηγική 2020, την οποία αναφέρετε και είπατε ότι θα πρέπει να την επανεξετάσουμε, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία παραμένουν. Παραδείγματο χάρη ο αριθμό των πτυχιούχων που έχουμε στην Ευρώπη σε σχέση με το τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν κάποια αυξητικές ε, τάσεις. Ε, υπάρχει επίσης η όλη συζήτηση αυτού του διτού δρόμου, αλλά κατά την άποψή μου αν ναι, ακολουθούμε μια τέτοια λογική, το να προσέχουμε λίγο και την ε, ε, διασπορά και την εγκατάλειψη του σχολείου, κυρίως σε επίπεδο μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι υπάρχει και διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος ε, πρωτίστως πλέον είναι σε θέμα ανθρωπίνων πόρων και κατάλληλης κατάρτισης. Θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση λοιπόν. Από την παρέμβασή σας ε, είδα ότι σταθήκατε στις προτεραιότητες που θέλετε να ακολουθήσετε, κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης και μέσω των συστάσεων φυσικά που θα μπορέσετε να προωθήσετε και εμείς σας ζητούμε να κάνετε και συστάσεις. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μου επιτρέπετε να επισημάνω κι εγώ, διότι αν όντω σήμερα η απασχόληση είναι η βασική κατεπίγουσα ανάγκη μας, ε, είπατε κι εσείς ότι δεν είναι μόνο η αποσχολησιμότητα αυτή η οποία θα πρέπει να μας ε, απασχολεί όταν ε, συζητάτε το θέμα της απασχόλησης και της παιδείας. Ναι, υπάρχει μια ανάγκη, αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο άτομα γενικότερης παιδείας και κατάρτισης και θα έπρεπε ίσως να αναφερθούμε και στη διαδικασία μετά το Παρίσι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι όσον αφορά την επικοινωνία Εάν σταθούμε πάρα πολύ στην ασφάλεια, ε, μπορεί η παιδεία να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Και επίσης θεωρώ ότι ίσως αν δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία και όσον αφορά ε, το πόσο σχετικά αντιμετωπίζονται κάποια θέματα στον πολιτισμό μας. Ε, για παράδειγμα, το να αναφερόμαστε σε κοινωνικές και δημοκρατικές αξίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να είναι και κοινέ αυτές οι αξίες. Επομένως, υπάρχει και ένα θέμα συνέχειας και ουσίας στα όσα προτείνουμε και εδώ θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη ε, παρατήρηση για να σκεφτούμε το όλο σχολικό σύστημα στο σύστημα της ανώτατης παιδείας και στα πανεπιστήμια θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να τυποποιήσουμε κάποιες πτυχές, την ε, ισοδυναμία για παράδειγμα και τη συμβατότητα των ε, ε, προγραμμάτων σπουδών, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να συγκρίνουμε, αλλά συμφωνώ ε, ε, νομίζω και μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και να γίνεται και κατάλληλη σύγκριση σε σχέση με σπουδαστές που έρχονται από όλες χώρες και όλη η συζήτηση είναι και στοιχείο ποιότητας και είναι πολύ σημαντική και επισήμανση που κάνατε για τα πανεπιστήμια του σήμερα. Εσείς αναφέρεστε κυρίως στα συστήματα τα οποία εφαρμόζονται στις Ηνωμένε Πολιτείε ή και σε άλλες χώρες για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της διδασκαλίας και της ευρωπαϊκής παράδοσης, ε, ε, η ευρωπαϊκή παράδοση που δεν είναι βέβαια ταυτόσιμη σε όλα τα σημεία, σχετίζεται με συνδυασμό και έρευνας ε, και αναζήτησης δεδομένων και πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη γιατί αλλιώς δεν προχωρούμε σε πολιτιστικά ζητήματα. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μόρκανο. Και τώρα ο κύριο Λέκοφ και με αυτόν ολοκληρώνεται η παρεμβάση. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με το ρητό ε, νους υγιής εν σώματι υγιή. Δεν είπατε τίποτα για τον αθλητισμό σήμερα. Ε, στην ακρόαση, στη διάρκεια της, ε, ε της ακρόασης σας το φθηνό είχατε πει ότι θα προωθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές και θα ενισχύσετε τις επενδύσεις σε ε, αθλητικές εγκαταστάσεις. Είπατε επίση ότι θα διατεθούν κονδύλια ύψου 300 εκατομμυρίων για τον αθλητισμό και ότι θα διοργανώνατε και μια εβδομάδα αθλητισμού για πρώτη φορά το φθινόπωρο. Και θα ήθελα να σας ε, τονίσω το σκάνδαλο της FIFA με τη σύλληψη 14 αξιωματούχων του συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτό θα επηρεάσει και του, τις μεγάλες, ε, τους μεγάλους συλλόγους αλλά και τους ερασιτεχνικούς συλλόγους του ποδοσφαίρου και είναι σημαντικό διότι αυτοί οι σύλλογοι, οι ερασιτεχνικοί ε, συμβάλλουν στην συμφιλίωση των ε, λαών και είναι σημαντικό ε, το Erasmus Plus να ενισχύσει και τα αθλητικά ιδεώδη και αυτό αφορά και το ζήτημα του μαζικού αθλητισμού. Η αξιολόγηση του πρώτου έτους απέδειξε ότι οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λαϊκού αθλητισμού και που ε, συμβάλλουν σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ λίγες. Πώς εσείς λοιπόν εσείς θα ενισχύσετε τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τι σκοπεύετε να κάνετε. Άλλο ερώτημα που σχετίζεται και με άλλα προγράμματα, όχι μόνο με το συγκεκριμένο. Υπάρχει πάντοτε μια σαφής ε, προτίμηση που επιδεικνύεται απέναντι στα μεγάλα έργα. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς τη δική σας γνώμη και να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του αθλητισμού. Θα ήθελα να συνοψίσετε σας παρακαλώ την άποψή σας για τον αθλητισμό, διότι όταν μιλούμε για τον πολιτισμό, όπως, είπα και νωρίτερα, χρειαζόμαστε υγεία, ενσώματη υγεία. Ευχαριστώ. Νομίζω κύριε Επίτροπε ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα ετέθησαν εδώ σήμερα, τα έθιξαν οι συνάδελφοι και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά τους νομίζω ότι το θέμα του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό, διότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στο, Συμβούλιο, στο Στρασβούργο ενέκρινε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα. Είναι και το θέμα του αθλητισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του θεματολογίου σας και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο θα μπορούσε να είναι ε, και μια πολύ σημαντική ένδειξη να συζητηθεί το θέμα και εν ώψη της Εβδομάδας Αθλητισμού το Σεπτέμβριο. Εμείς θα κάνουμε και μια σχετική ακρόταση ή μια πρόταση μάλλον για ακρόαση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα να κυρώσουν και τις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και ίσως και η ίδια Ευρώπη θα μπορούσε να υπογράψει, δεδομένου ότι νομικός έχει αυτή τη δυνατότητα και η ίδια ω Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση. Σα δίνω το λόγο λοιπόν για τι επόμενε απαντήσει. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετά το Παρίσι, post-Paris process, ε, συνεργαζόμαστε με τους Υπουργούς Παιδείας σε αυτές τις χώρες στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργαζόμαστε με υφυπουργεία ή αρμοδίους υπουργού σε περιφερειακό επίπεδο γιατί η αρμοδιότητα της παιδείας είναι αποκλειστικά και μόνο στα χέρια της περιφέρειας. Το ίδιο στη Γερμανία είναι ε, υπουργό ομοσπονδιακού κρατηδίου. Ε, κρατηδίου αυτός που έχει την ε, αρμοδιότητα για την παιδεία. Στη Γαλλία και σε άλλες χώρες συνεργαζόμαστε με τον Εθνικό Υπουργό Παιδείας αναλόγως με το που, ποιος τομέας έχει την αρμοδιότητα για την παιδεία. Τώρα, προς τις μειονοτικές γλώσσες είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Πρέπει να βρούμε μια καλή λύση και για τα θέματα copyright, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν έχει μόνο να κάνει με τις νομικές ε, διαστάσεις του θέματος αυτό, έχει να κάνει και με τον πολιτισμό οι μικρές γλώσσες, οι μειονοτικές γλώσσες, ο σεβασμός των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καυτό θέμα ε, στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Είμαι αισιόδοξο. Διότι ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο εσθονός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μιλάει εσθονικά, τα οποία δεν είναι και η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ευαίσθητος σε σχέση με το γλωσσικό ζήτημα. Όμως, πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, γιατί η ενιαία ψηφιακή αγορά δεν θα πρέπει να σημαίνει την κατάργηση του σεβασμού και της χρήσης των μικρών ή μειονοτικών γλωσσών επίσης. Κυρία Ward, βεβαίως συμφωνώ απολύτως μαζί σας για το ρόλο και τη σφινισφορά των μεταναστών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα ε, μάλλον. Ε, η συζήτηση που έγινε πρόσφατα δεν έγινε για τη συνεισφορά των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ε, ε, έχει κυρίως να κάνει με θέματα ασφαλείας. Και μπορούμε να συζητούμε επί μακρόν για τη συνεισφορά των μεταναστών η οποία βεβαίως και ισχύει στην ευρωπαϊκή κουλτούρα όμως προς το παρόν το κύμα μεταναστών δημιουργεί θέματα ασφαλείας και αυτά δεν άπτονται της πολιτικής κουλτούρας και πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει τη δική της πρόταση για τη μεταναστευτική πολιτική και στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ρόλο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών υπάρχουν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, όπως υπάρχουν και πολλά στοιχεία για τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου και για τη συνεισφορά του διαλόγου αυτού στην κοινωνική ένταξη και στη σταθερή κοινωνία. Ο διαπολιτισμικός διάλογος παίζει ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό και κατά τη δική μου άποψη και γι' αυτό συναντήθηκα με οργανώσεις νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σας αναφέρω ότι ε, με πολλές και διαφορετικές οργανώσεις νέων, όχι μόνο πολιτικές αλλά και πολιτισμικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και άλλες και κάθε φορά που πηγαίνω σε κάποιο κράτος μέλος, όποιο και αν είναι αυτό, προσπαθώ να επισκεφθώ ένα κέντρο κοινότητα, σε κοινοτικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, ένα κέντρο νεότητας να δω πώς προωθούν το διαπολιτισμικό διάλογο με συγκεκριμένα σχέδια, προγράμματα, έργα και πώς προωθούν την κοινωνική ένταξη ή την κοινωνική επανένταξη. Κύριε Μοργάνο, να σας πω επίσης ότι η εκπαίδευση δεν έχει μόνο να κάνει με την απασχολησιμότητα βεβαίως και γι' αυτό στηρίζω την ιδέα της δημοκρατικής αγωγής του πολίτη, της δημοκρατικής ηθαγένειας. Βασικός στόχος των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι να εκπαιδεύουν πολίτες δημοκράτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες, τα ε, τους θεσμούς, τους, ε, τα δικαιώματα ενός πολίτη σε μια δημοκρατία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η διαδικασία μετά το Παρίσι και ο ρόλος της εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια. Και μάλιστα η διάσταση της ασφάλειας υπερεκπροσωπείται αυτή τη στιγμή κατά πάσα πιθανότητα λόγω ε, της ε, δυσκολίας της κατάστασης, του, της ευθραυστότητας αν θέλετε της κατάστασης. Ωστόσο, ε, βασικό μέλημα της εκπαίδευσης για μένα είναι να εκπαιδεύει δημοκράτες, πολίτες. Κύριε Νέκοφ, έχετε δίκιο. Δεν αναφέρθηκα σε λεπτομέρειες στο θέμα αυτό. Ε, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε λεπτομερή συζήτηση για τα αθλήματα και τον αθλητισμό εδώ στην Επιτροπή. Πράγματι, 300 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν στο πλαίσιο του Ερασμού ΣΥΝ για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού σε επίπεδο κοινότητας, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέτος, χάρη στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, θα έχουμε την δεύτερη σχετική συνάντηση ε, για τον αθλητισμό, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Πιστεύω ακραδάντως σε αυτό τον ρόλο κοινωνικοποίησης που παίζουν τα αθλήματα και ο αθλητισμός γενικότερα, γιατί τα θετικά πρότυπα είναι απαραίτητα στις τοπικές κοινωνίες για να προσελκυστούν στην κοινωνία, στον κορμό της κοινωνίας οι αλωτριωμένοι ή αποξενωμένοι. Είναι ο βασικός παράγοντας κοινωνικοποίησης αυτός. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Άλλωστε ο αθλητισμός για μένα έχει να κάνει με ε, το χτίσιμο του, της αίσθηση της κοινότητας, του ανήκει σε μια κοινότητα. Στηρίζω πολύ το στον αθλητισμό και η θέση μου για τη FIFA αν, ε, δεν ξέρω αν είδατε την Τρίτη το βράδυ στο Στρασβούργο της περασμένης εβδομάδας έκανα μια δήλωση για τη FIFA γιατί είχε μπει αυτό το θέμα στη μερίσια διάταξη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως γνωρίζετε υιοθέτησε ε, ψήφισμα γι' αυτό. Τώρα για τα project μεγάλου βεληνικού και μικρού βεληνικού μπορούμε να το συζητήσουμε το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Νομίζω ότι σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μέρα μας. Ε, σας ευχαριστώ και για τις αφέστατες απαντήσεις σας και ε, από εκεί και πέρα και για τη στοιχεία που μας δώσετε που θα συζητήσουμε στην ε, συνεδριάση μας πιο αναλυτικά. Υπάρχει όμως ένα στεναρό μήνυμα το οποίο πρέπει να προκύψει από τη συζήτησή μας και ότι αυτό είναι ότι η πρόκληση για την Ευρώπη είναι ε, εκπαιδευτική και πολιτιστική και νομίζω ότι εσείς ε, θα εργαστείτε για να θέσετε τα θέματα αυτά στο επίκεντρο και να προβληθούν λίγο καλύτερα το θέμα της παιδείας, το θέμα του πολιτισμού, της δημιουργικότητας, των πολιτικών για την νεολαία και φυσικά των ε, δεσμεύσεων στον τομέα του αθλητισμού ως ε, βασικοί παράγοντες για να μπορέσουμε να υπερκεράσουμε αυτή την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόκληση δεν θα πρέπει να συζητούμε μόνο θέματα ασφάλειας ε, και θέματα απασχόλησης, όσο σημαντικά και να δεν θα πρέπει να χάσουμε και το στόχο αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ανάλυση σας. Δεύτερο σημείο, σας εφιστώ την προσοχή για τον προπολογισμό. Ε, εμείς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να διατηρήσει και να υπερασπιστεί τον προπολογισμό για το 2016, αλλά και να είστε ανοιχτοί και στα πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα υποβάλει η Επιτροπή Πολιτισμού, κύριε Επίτροπε,

και είναι πολύ σημαντικές ε, και οι πτυχές που λαμβάνει υπόψη της. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η πρωτοβουλία αυτών των συναντήσεων σε περιφερειακό επίπεδο για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να έχουμε επενδύσει ε, ε, μέσω του σχεδίου Juncker και συγκεκριμένε προτεραιότητε. Πιστεύω ότι πολλές χώρες και οι δικοί μου ασχολούνται με συγκεκριμένε πλατφόρμες για την παιδεία και τον πολιτισμό και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε και κάποιες ανταλλαγές απόψεων μαζί σα για να δούμε λίγο προ τα που οδεύουμε και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρουμε κι εμείς. Ελπίζω τουλάχιστον ότι από αυτού θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Σας χαιρετώ και επίσης να υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι τώρα έχουμε μια πολύ σημαντική ενημέρωση και κλεισμένων των θερών από την κυρία Καμερέβερτ για τον τριμερή διάλογο για τη στρατηγική για τις τηλεπικοινωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μείνετε, ε, μόνο όσοι δικαιούστε φυσικά να μείνετε στις συνεδρίες και κλεισμένων των θερών. Ε, σας χαιρετώ και θα συναντηθούμε στις 2.30 αν δεν κάνω λάθος για να ε, επισκεφθούμε τον οργανισμό ΕΑΤΣΕ.